Απορρίπτεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 379 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 379. Πέρας. Απορρίπτεται. «380 υπέρ». Κατά. Αποχές Αποδεκτεί. «381 υπέρ». Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. «381 ελέγχουμε». Πέρας. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. 383 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 402 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 403 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 404 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 406 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 408 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 410 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 411 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 413 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 414 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτής. 16α 417 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 431 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 449 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Check 449 I close the vote. Rejected. Rejected. Λοιπόν, απορρίπτε, απορρίπτεται Θεούλη μου. 4.50 υπέρ, κατά, αποχές. Και αυτό χρειάζεται έλεγχο και πάλι. 4.50. Ένα EPP. Ένας υπεράριθμος εξακολουθεί να είναι από το ΑΕΛ, ζητώ συγγνώμη. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.55 υπέρ. Κατά. Uh, 4.55. 4.55 και αυτό το ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 456 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 454 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. 4.51 μέχρι και 53. Είναι τρεις τροπολογίες υπέρ. 51, 52, 53. Κατά αποχές εγκρίνονται. 4.57 υπέρ. Κατά. Πάλι έλεγχος παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίψετε. 4.64 ε, υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. 4,50, συγγνώμη, 4,64. Πέρας. Απορρίπτεται. 4,58 είπε. Κατά. Έλεγχος. 4,58. Παληθεύουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 4.59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.65 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.62 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 4.62 Πέρας. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 460 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μάλλον, αλλά στην ελέγξουμε την 460. Πέρας. 463 υπέρ, απερίφθη προηγούμενη, κατά αγωγές απορρίπτεται, 466 υπέρ, κατά αποχές δεν είμαι βέβαιος, 466 ας την ελέγξουμε παρακαλώ, πέρας, απερίφθη, μάλιστα. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 478 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Α, όχι, όχι, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Απερίφθη σαφέστατα. Η 478 απερίφθη. Αν θέλετε να την ελέγξουμε, ήταν σαφέ δικό μου λάθο, λέει ο πρόεδρο. Ε, συμβαστική 19 υπέρ Πώς ξέρετε ότι έχει αλκοόλ αυτό που πίνω μέσα. Το νερό. Compromise 19 in favor. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 484 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 485 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 496 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 500 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ορίστε 500 υπέρ κατά Ας το αλλάξουμε καλά. Έχετε απολύτως δίκιο, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται 501 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε και αυτή. Πέρας. Απορρίπτεται επίσης. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Συμβαστική 28. Πέρασε ψηφοφορίες. Ισοψηφία απορρίπτεται. Η τροπολογία 500 Δύο λέει ο πρόεδρος. Μαζί με την 3, 4 και 5. Όλες μαζί αυτές. Γιατί ταυτίζονται. 502, 503, 504, 505. Κατά. Η συμβιβαστική 28 απερίφθη λόγω ισοψηφίας. Και εφόσον απερίφθη ψηφίζονται δυστυχώ οι τροπολογίε αυτές διότι δεν καλύπτονται άρα συν μία ώρα ψηφοφορίες. Αν το πάτε έτσι. Λοιπόν, τέσσερις τροπολογίες ομού. 502 και 5 Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρασε εγκρίνονται. Οπότε τώρα μπορούμε να πάμε στην τροπολογία 520. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. I close the vote. Πέρας. 521 ε, υπέρ. Κατά. Έλεγχος και πάλι χρειάζεται. Δεν ψηφίζεται όλοι μάλλον. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 530 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 530 λήξεις εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 536 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται 537 υπέρ όχι όχι 5.41 πάμε υπέρ, κατά, δεν ξέρουμε τι έγινε τώρα, 5.41 έλεγχος. Check the amendment, I close the vote. Rejected. Rejected. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 544, το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 552 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 557 το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 557 το τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 565 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 566 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 573 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 589 υπέρ κατά α, εγκρίνεται τσεκ, καλά ελέγχουμε λοιπόν τι ψηφίζουμε την 589 πέρασε κρίθηκε. συμβιβαστική α υπέρ κατά από 23 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 23. Η συμβαστική α εγκρίθηκε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική σ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική δ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 και 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές τι έγινε α όχι έχει, καταπέσει δεν ψηφίζουμε την 69 εφόσον εγκρίθηκε 68 συμβιβαστική G από την 68 πάμε στη G συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 85 και 87 μαζί υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε αυτό τις δύο αυτές τροπολογίες 85 και 87 πέρας. μισοψηφοί απορρίπτονται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες έχουμε τώρα. 103, 104 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 105 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 105. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα ήταν αυτό. Τροπολογία 1. Υπέρ. Αν μπλοκ λέει ο κύριος Λάγκεν, όχι απαντάνε. Ε, τροπολογία 1. Με τη σειρά θα τις ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Οι 2. Υπέρ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 Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται ολόκληρη η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Λάγκεν. Εύκολη δεν ήτανε. Μια ώρα ψηφοφορία σχεδόν. Φαντάζομαι πόσες ώρες ήταν η προετοιμασία για τις ε, Μπορεί να ήταν και 100 ώρες. Σας ευχαριστώ όλους σας και τους και ηγητές Επίσης, όχι μόνο τον εισηγητή τον ίδιο, όλους σας που κάνετε τόσο σκληρή δουλειά για τις συμβαστικές τροπολογίες και όλους τους σκιώδεις επαναλαμβάνω. Πάμε στο επόμενο θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι του κυρίου, του κυρίου Ταμπουράνο, του Ντάριο Ταμπουράνο. Σήμανση αποτελεσματικότητα ενεργειακής απόδοσης και ανάκληση οδηγίας του 2010. Μια να λοιπόν. Πρώτη συμβαστική. Όχι, μαζί. Let us start. Let us start then. Ωραία, λοιπόν, ξεκινούμε. Δύο συμβαστικές. Η υπαριθμών 1 και η R4α μαζί. Υπέρ. Τα τα. Αποχές. Αποδεκτές. Αρχικό. Όχι. Προσθήκη ε, στο, στη συμφαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απερίφθη. Προσθήκη 2. μαζί με δύο τροπολογίες 314 και 365 υπερθυμών 2 προσθήκη υπέρ κατά επαληθεύουμε. Πολύ σημαντικό. Και επαληθεύουμε. Δύο τροπολογίες στην προσθήκη 2 και πέρα στις ε, ψηφοφορίες επερίφθησαν και πάμε. Στην 317 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 16 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απερίφθη 338 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 366 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Συμβαστική 3α παρακαλώ υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. Προσθήκη παριθμών 1 στην συμβαστική 3α υπέρ κατά επαληθεύουμε. Λοιπόν, προσθήκη 1 ε, στην 3α συμβιβαστική. Απερίφθη. 3β συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση. Επαναλαμβάνω την ερώτηση για να ρωτήσω αν έχετε κάποια ένσταση στην ε, ψηφοφορία της ε, ε, τροπολογίας αυτής, της προφορικής. Ο κύριος τουρμέ, ναι, εμείς. Και λυπούμε. Τέσσερις πρέπει. Να είμαστε. Καλά, λοιπόν, δεν ψηφίζεται η προφορική. Προσθήκη 1 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 4. Και γυρνάμε τις σελίδες. Συμβαστική 4 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4, 5, 2 υπέρ. Επαληθεύουμε. 452 λοιπόν. Πέρας. Και απερίφθη. 465 υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε. 465 πέρας. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη παριθμών 1 στη συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Προσθήκη 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 495 με την προσθήκη 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε πολλές σελίδε και πάμε στη συμβαστική 8. Με τη σελίδα υπαριθμών 56 για όποιον έχει έγγραφο στα χέρια του. Τι να ψηφίσουμε τώρα. Την προσθήκη παριθμών 1 στη συμβαστική 8. Επαλήθευση. Όχι, όχι. Συμβαστική 7. Θα ακολουθήσει η 8. Πρώτα την 7. Επαλήθευση. Dear Αγαπητοί φίλοι, ένα, ένα λεπτό, ένα λεπτό, με ηρεμία. Σελίδα 42. Ένα λεπτό. Είχαμε ψηφίσει μέχρι πριν από τη συμβαστική 8 την προσθήκη για τη συμβαστική 7 της σελίδας 42. Και από ό,τι αντελήφθη ζητήσατε επαλήθευση της ψηφοφορίας αυτής, δηλαδή σελίδα 42. Παρακαλώ αγαπητοί φίλοι. Προσθήκη στην 7, συμβιβαστική. Παρακαλώ, βρείτε το, βρείτε το ήρεμα ήρεμα προσθήκη στην συμβιβαστική 7 αριθμός προσθήκης 1 μια και είναι διαφορετικές σελίδες ανάλογα με την περίπτωση οπότε καταλαβαίνω ξανά ε, λέω την προσθήκη της συμβιβαστικής 7 και άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει, το καταλάβατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Και να κρίθει. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Επαληθεύω. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, προσθήκη παριθμών 1 τώρα για τη συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε. Πέρασε στις προφορίες εγκρίνεται και άρα προχωρούμε στην προσθήκη 2. Προσθήκη 2 της συμβαστικής 8. Τα λέω έτσι γιατί έχουμε διαφορετικές σελίδες. Υπέρ, κατά, επαληθεύουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. Προσθήκη 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Εξακόσια δεκαπέντε υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε 615 πέρας 619 Είπε, κατά 609 συγγνώμη αποχές και επαληθεύουμε 609 πέρας και εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη υπερθμών 1 στην συμβαστική 9 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. Προσθήκη υπερθμών 1 στη συμβαστική 9 και απερίφθη. Προσθήκη 2 Στη συμβαστική εννέα υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε. Πέρας. Και απερίφθη. Ε, προσθήκη τρία Υπέρ. Κατά. Εποχές και απερίφθη. Προσθήκη 4 στη συμβαστική 9 υπέρ κατά απερίφθη. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 128 Επαληθεύουμε λοιπόν και πέρασε προφορία Απερίφθη. 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 629 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 631 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε 631 Πέρας. Και απερίφθη. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 635 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 είπε μάλλον 100 εννοεί, 358 μαζί υπέρ, κατά αποχές απερίφθησαν. Όχι, επαληθεύουμε. 100 και 358 μαζί. 100 και 358. Πέρας. Απερίφθησαν. 638. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα, 638. Πέρασε. Εξακόσια υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 646 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 659 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ε, προσθήκη 5β υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε. 5β προσθήκη. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. 517. Προσθήκη 6. Υπερ κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική, συμβαστικό παράρτημα υπέρ κατά αν πέρας Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη 685 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 1 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβαστική R2, ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ρο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική ρο 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρο 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρο 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ρο 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ρο 11α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρο 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ρο 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρο 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ρο 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ρο 15α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ρο 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, προσθήκη υπέρ, κατά. Για να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Άποχες απεριεύθη. Ρο 17. Συμβαστική ρο 17 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 23. Έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί. Σας ενημερώνω και πάμε στη 285 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το επαληθεύσουμε. Πέρας. 286 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε τη 286. Πέρας. Απέρευτη συμβαστική ρο 19 υπέρ κατά. Αποχές επαληθεύουμε και πάλι. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Ρο 20 συμβαστική, ρο 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Βλέπετε το ρόφημά μου και ζηλεύεται από ό,τι βλέπω. Το καταλαβαίνω, κατανοητών. Ρο 20α συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. Ρο 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία και πολύ σημαντική. Ηλεκτρονικές τρεις στον αριθμό. Σύνολο των τροπολογιών που εγκρίθηκαν είναι η πρώτη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Τώρα, σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 63 ψήφους. Υπέρ. Καμία ψήφο. Κατά και καμία αποχή. Κύριο Στουρμέζα δικαστικό. Πρόεδρε, θέλω πριν προχωρήσουμε στην απόφαση για το πώς θα ψηφίσουμε ως προς την εντολή, θέλω ενός λεπτού διακοπή. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Δύο λεπτά διακοπή. It will be one voting. Μία ψηφοφορία. If, if not,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 για τις ε, διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι, ένα λεπτό. Θα πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Ήτρε έχουμε 67 πλήρη μέλη. Το 50% είναι 33,5. Χρειαζόμαστε 34 υπέρ. Για υπέρ, γιατί θα πρέπει να έχουμε την πλειοψηφία όλων των μελών της Επιτροπής ΙΤΡΕ, όχι μόνο τους παρόντες. Αλλά αυτό δεν αφορά τους α, αναπληρωτές. Μόνο τα πλήρη μέλη. Αυτό είναι ο κανονισμός και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Γιατί το θέμα θα πάει στην Ολομέλεια. Δηλαδή δεν είναι ε, εντολή για διαπραγμάτευση στον ε, τριμερή διάλογο, γιατί ξέρετε ότι στην πρόταση νομοθετικού περιεχομένου είχαμε 66 ή 67 έναντι κανενός. Γι' αυτό θα πρέπει να πάμε στην ε, Ολομέλεια την πρόταση. Δεν πάμε απευθεία στον τριμερή διάλογο. Σας ευχαριστώ τελευταία έκθεση Προϋπολογισμός 2017 εντολή για τον τριμερή διάλογο. Θα πρέπει να τελειώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 4 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές αποδεκτή. Τροπολογία 8, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 8 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3α υπέρ, κατά, αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ 24 συγγνώμη ε, αποδεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 28 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 28 παρακαλώ πέρας απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή 36 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 38 υπέρ, κατά αποχές αποδεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ, η οποία και άρχεται. Πέρας. 51 υπέρ, κατά 9. Ε, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ και να συγχαρούμε τον εισηγητή, δηλαδή τον υποφαινόμενο. Αυτό περίμενα. Αυτό περίμενα. Δεν με εκπλήσει καθόλου η αντίδρασή σας. It's me, it's me, Προχωράμε λοιπόν τώρα στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας. Έχουμε τέσσερις εκθέσεις. Ε, θα ήθελα να τελειώνετε με τις συζητήσεις σας ε, γύρω από το γύρω από το συντονιστή, κύριε Κάρινς. Αν θέλετε μπορείτε να αποχωρήσετε, θα μας διευκολύνατε. και όλοι από το ΕΛΚ που, που φαίνεται ότι θέλουν να αποχωρήσουν. Αγαπητοί φίλοι και σύμβουλοι του ΕΛΚ, παρακαλώ απομακρυνθείτε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το πακέτο της κυκλικής οικονομίας Έχουμε τέσσερα νομοθετικά κείμενα και τους εισηγητές και τους σκιώδεις για κάθε έκθεση. Έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας, ίσως ε, υπερβούμε κατά 10 λεπτά και ζητούμε συγγνώμη από τους διερμηνείς εκ των προτέρων, εάν τελειώσουμε στην μία παρά 20. αλλά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε τέσσερις προτάσεις της Επιτροπής, τρεις εισηγητές και, τρεις εισηγητές, με συγχωρείτε, και πολλούς σκιώδεις. Έχουμε 21 σκιώδεις, γι' αυτό καθένας θα πρέπει να αρκεστεί στο 1,5 λεπτό. Σας παρακαλώ. Αρχικά θα έχουμε τρεις εισηγητές. Ο κύριος Φέντερλει αντικαθιστά τον κύριο Τελίτσκα. Ο κύριος Φέντερλει θα μας παρουσιάσει δύο εκθέσεις. Και ο κύριος Πόχε και Φερέιρα θα είναι οι επόμενοι ομιλητές και θα μιλήσουμε ο καθένας για μία έκθεση. Ο κύριος Φέντερλεϊ λοιπόν έχει το λόγο για 7-8 λεπτά για να έχουν και άλλοι τη δυνατότητα να μιλήσουν. Κύριε Φέτελε, έχετε να μιλήσετε για δύο θέματα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ο κύριος ε, Τελίτσκα ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Είχαμε μία καρποφόρα συζήτηση με τον κύριο Τελίτσκα. Μιλήσαμε για τις ε, ηλεκτρονικές στήλες. Ε, μας λέει λοιπόν ότι θα σας μιλήσω για τις ηλεκτρικές στήλες και τους ορευτές και τα απόβληκά τους. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να σας ε, παράσω ένα κείμενο για όλα αυτά τα θέματα που θα απασχολήσει την Επιτροπή. Στόχος είναι να θίξουμε ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται ή καλύπτονται ε, ανεπαρκώς από την πρόταση της Επιτροπής για να υπάρχει και συνεκτικότητα. Ως προς το πακέτο αποβλήτων η νομοθεσία είναι περίπλοκη. Η κυκλική οικονομία είναι συνώνυμη με τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ο κύριος Τελίτσκα ε, έχει μία ολιστική προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μία νέα οικονομία, αν βρούμε τα σωστά κίνητρα και ε, μία εξισορρόπηση. Πολλές φορές μιλάμε για τα σωστά κίνητρα έτσι ώστε η διαχείριση αποβλήτων να είναι σωστή. Αλλά τα, αυτά τα κίνητρα δεν υπάρχουν στην πρόταση της Κομισιόν. Γι' αυτό ο κύριος Τελίσκα έχει επανεισαγάγει οικονομικά και άλλα κίνητρα στην πρώτη πρόταση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη για να φτάσουμε στο στόχο ως προς την διαχείριση των αποβλήτων. Πρόκειται για ένα παράρτημα στις τρεις οδηγίες και θα ενισχυθεί και σε άλλες οδηγίες. Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ε, συλλογή αποβλήτων και γι' αυτό θεωρεί ο κύριος Τελίτσκα ότι θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή διαχείριση των αποβλήτων προς ανακύκλωση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτές τις προδιαγραφές που είναι υποχρεωτικές για ορισμένα κράτη-μέλη, που να είναι υποχρεωτικές για όλα τα κράτη-μέλη, για να υπάρχουν ίση όροι πρόσβαση στην αγορά και ίση διαχείριση ο κύριος Τελίτσκα θα ήθελε να θίξει και ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τον όλο ε, κύκλο. Ε, δεν μιλάμε για, την, ε, για τις φορτωτικές και αποστολές των αποβλήτων. Εάν μιλάμε για ενδοκινοτική διαχείριση θα πρέπει να βρούμε πιο σωστά συστήματα χωρίς να υπάρχει διοικητικό άχθος. Έχει μεγάλη σημασία η σωστή διαχείριση, γι' αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη κάτι την αναθεώρηση της οδηγίας για την αποστολή ή φόρτωση των αποβλήτων. Έχει λοιπόν σημασία να λάβουμε υπόψη την νομοθεσία για καλύτερη διαχείριση και νομοθέτηση κατά την ε, διαχείριση των αποβλήτων του πακέτου. Επίσης να δώσουμε πληροφορίες για τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τη συμβίωση με τη βιομηχανία για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Τώρα, σε σχέση με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, ο κύριος Τελίτσκα λέει τα εξής. Μία από τις πολλές προτάσεις σχετίζεται με μία πλατφόρμα επικοινωνίας για να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και διαφόρων τομέων, λαμβάνοντας υπόψη και την βιομηχανία αποβλήτων. Θα πρέπει λοιπόν η πλατφόρμα επικοινωνίας να μας οδηγήσει σε μια καλύτερη επίβλεψη των, ε, της διάθεσης χώρων και χωρητικότητας. Επίσης, ο οικονομικός τομέας βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να δει κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε έναν στόχο για την υγειονομική ταφή ανά χιλιόγραμμο, ανά άτομο κατέτος, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο προ... πρόληψης και πρόβλεψης. Έτσι θα μειώναμε τα συνολικά απόβλητα που παράγονται ετησίως. Επίσης θα ήθελε να, υποστηρίξει, την υποχρεωτική, τον υποχρεωτικό διαχωρισμό των βιοαποβλήτων, αλλά αυτό το θα το δούμε γενικότερα στον κανονισμό περί αποβλήτων. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ήθελε να θίξει ο κύριος Τελίτσκα, αλλά ε, γενικά θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ολοκληρωτική προσέγγιση και ο κύριος Τελίσκα ζητεί συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε για την παρουσίαση αυτών των δύο ζητημάτων. Και τώρα θα μιλήσει ο κύριος Μυροσλάβ Πόχε σε σχέση με την τροποποίηση της οδηγίας 2008 κάθετος 98 για τα απόβλητα. Ευχαριστώ πολύ. Η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει χρήματα από ε, τα απόβλητα τα οποία είναι πόροι. Και όχι μόνο χάνουμε χρήματα, αλλά βλάπτουμε και το περιβάλλον. Πρώτες ύλες πόροι λοιπόν που δεν ανανεώνονται ε, είναι τα απόβλητα, πολλά από αυτά και χρειάζεται να έχουμε μια νέα οικονομία, μια κυκλική οικονομία για να κάνουμε ε, οικονομία να μην βλάπτουμε το περιβάλλον και να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. 2,5 δισεκατομμύρια τόνους αποβλήτων παράγουμε. Ε, άρα το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας δεν αρκεί. Υπάρχει θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητεί ε, πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Γι' αυτό προτείνω εγώ αυτούς τους πιο φιλόδοξους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, είναι στο ύψος των περιστάσεων και αυτά που προτείνει δεν πρόκειται να μειώσουν τα απόβλητα στις χωματερές ε, ούτε τα απόβλητα που αποτεφρώνονται. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτής της οδηγίας. Οι ορισμοί θα πρέπει φυσικά να είναι τελείως ξεκάθαροι και χωρίς αφησιμίες και πιο εναρμονημένοι. Το θέμα δεν είναι μόνο τα αστικά απόβλητα, ε, αλλά και ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση συνολικά των αποβλήτων. Προτείνω λοιπόν ένα νέο ορισμό ε, των εμπορικών και οικονομικών και μάλλον συγγνώμη, βιομηχανικών αποβλήτων. Και μετά υπάρχουν και τα υπολείμματα τροφίμων και τα απόβλητα από ε, τρόφιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας στη ε, Γεωργία. Οι παράνομες χωματερές είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό επίσης το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η ε, ευθύνη των παραγωγών είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει για να δούμε πώς διαχειρίζονται αυτά τα απόβλητα. Λοιπόν, είναι μια προσέγγιση συνολική και θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι και οι γεωργοί και οι εκτινοτρόφοι. Ε, λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι ενίσχυση των στόχων. Ε, δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης δεν καλύπτει πάρα πολλά ε, σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση των λέων που πρέπει να φτάνει το 60% και μέχρι το 2030 ακόμα περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ασαφής. Εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται με το μέθοδο υπολογισμού. Πώς υπολογίζεται ε, κάθε φορά ποιο πράγμα πρέπει να το ξέρουμε για να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Χρειάζεται νέα μέθοδος που μην αφορά αποκλειστικά τις ποσότητες αλλά και την παραγωγή και γενικότερα στοιχεία και την κατακεφαλή παραγωγή απορριμμάτων και αποβλήτων. Δεν έχουμε καλές αναλύσεις και δεν μπορούμε να αξιολογούμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων κάθε φορά. Γι' αυτό θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε τουλάχιστον, να μας κάνει μια τέτοια ανάλυση. Επίσης, άλλο ε, θέμα είναι η προστασία των καταναλωτών και πάλι δεν καλύπτεται παρκώς από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να φτάσουμε στους επιθυμητούς στόχους και ε, η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων είναι να μειώνεται στην πηγή, η παραγωγή τους δηλαδή. Ευχαριστώ τους και ηγητές και ελπίζω σε μελλοντικές συνεδριάσεις να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς φιλόδοξους για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε στην ε, προστασία του περιβάλλοντος και να εκμεταλλευτούμε τους πόρους που είναι τα σκουπίδια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, που παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Και τώρα, που έχει να κάνει με τα απόβλητα και ε, τις συσκευασίε. Ο κύριος Φερέιρα είναι εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς, ε, θέλω να πω κάτι γενικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας προτείνει ε, διάφορα πράγματα για τις συσκευασίε και τα απορρίμματα συσκευασία και φρονεί ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο κάτω για τη χρήση των αποβλήτων αυτών και την επαναχρησιμοποίησή του. Αυτό θα έχει πλέον εκτήματα και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πρώτη ύλη, σε πόρο, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια κυκλική οικονομία στο βαθμό του δυνατού στο βαθμό του δυνατού γιατί η ανακύκλωση έχει σημαντικά πλέον εκτήματα ως προς την επαναχρησιμοποίηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται το Υπάρχουν προϊόντα που έχουν περιορισμένο κύκλο ζωής. Δεν είναι πάντα τέλειος ο κύκλος ε, και η επαναχρησιμοποίηση δεν ε, είναι κάτι που αφορά όλα τα απόβλητα. Όσο καλή ε, προσέγγιση και να έχει κανείς. Γενικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνει τους στόχους ε, της ε, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Είναι πιο φιλόδοξη σε σχέση με το παρελθόν, ειδικά για συγκεκριμένα υλικά στις συσκευασίες και προβλέπει και νέους κανόνες για τον υπολογισμό ε, για το πώς γίνονται σεβαστοί οι στόχοι. Εναρμονισμένους κανόνες επίσης για να δούμε πώς ε, θα αξιολογείται η τήρηση των στόχων. Η παρούσα πρόταση γνωμοδότηση συμφωνεί γενικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προσέγγιση και τους στόχους, αλλά προσθέτουμε και κάποια στοιχεία σημαντικά κατά την άποψή μας. θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν βρίσκονται στην ίδια φετηρία. Μπορεί να υπάρχουν κοινοί στόχοι, αλλά δεν κινούμε όλοι από το ίδιο σημείο. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταβάλει διαφορετική προσπάθεια, έτσι ώστε να φτάσει στους ε, καθορισμένους στόχους. Η πρόταση αναγνωρίζει ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν στήσει τις απαραίτητες ε, δομές διαχείρισης και υποδομές ακόμα, πράγμα που δυσκολεύει την κατάσταση. Εμείς δεν αφισβητούμε τους στόχους, αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας δεν ξεκινάει από το ίδιο σημείο, οπότε χρειάζεται προσωρινά κάποια ευελιξία για να μπορέσει η κάθε χώρα να προσαρμοστεί. Αυτή την ευελιξία προτείνουμε και την ελαστικότητα στο σχέδιο γνωμοδότησής μας. για να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης, παρέκκλησης, χρονικής επαναλαμβάνω, για τους νέους αυτούς στόχους. Εδώ υπάρχουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις. σταδιακή προσέγγιση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ε, καλή η σύγκληση και εναρμόνιση, αλλά χρειάζεται προοδευτική ε, προσαρμογή των χωρών που δεν είναι όλες στην ίδια μοίρα όλα αυτά προβλέπονται και ως έγκαιρη προειδοποίηση είναι μια νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να είναι οι συστάσεις προσαρμοσμένες στην κάθε πραγματικότητα, σε κάθε κράτος μέλος, για να γίνονται σεβαστές. Άλλο σημείο που ξαναβρίσκουμε στο σχέδιο νομοδότησης. Η διεύρυνση της ε, τη της ευθύνης του παραγωγού. Αυτό έχει να κάνει με την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. Να έχουμε συστήματα που να επιτρέπουν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση συσκευασιών, είτε προέρχονται από τον τελικό καταναλωτή, ε, είτε από κάποιον άλλο χρήστη. Αυτό έχει να κάνει με την ευθύνη του παραγωγού. Δηλαδή, πολλές φορές δεν επιλέγει ο τελικός χρήστης, ο τελικός καταναλωτής τη συσκευασία του προϊόντος. Ε, αυτή η έννοια της επέκτασης της ευθύνης του παραγωγού είναι κάτι που μας προβληματίζει. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη που πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Να δοθούν κίνητρα. Θα πρέπει η βιομηχανία να καταλαβαίνει ότι και οι συσκευασίες έχουν νόημα, ε, δηλαδή ότι είναι πόρος και θα πρέπει ε, να ασχολείται με αυτό ενεργά ο κάθε παραγωγός του προϊόντος. Δεν είναι κάτι το δευτερεύον η συσκευασία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Και παρακαλώ. Από την Ήτρε, κύριος εισηγητής και αναπληρωτής όποιος είναι, να λάβει ε, μετά τους σκιώδεις. Η κυρία Μποναφέ είναι υπεύθυνη και για τα τέσσερα θέματα ως κύρια στην ΕΝΒΗ. Ε, λοιπόν, μετά τους Σκιώδη θα σας παρακαλέσω κύριε Πονάφη, να λάβετε το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόιλ έχει το λόγο. ΕΛΚ. Ναι, ευχαριστώ. Στην έκθεση για την οδηγία για τις συσκευασιε υπαρχουν υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα που μας απασχολούν ακόμη και νομίζω ότι τα συστήματα διευρυμένης ευθύνη ε, του παραγωγού είναι καλά και φέρνουν αποτελέσματα, αλλά σε κάποια σημεία ίσως ε, δεν θα έπρεπε να παρέμβουμε. Καταρχάς, υπάρχει, στο, υπάρχει ο κανονισμός για τα απόβλητα, λειτουργεί, έχει φέρει συστήματα με αποτελέσματα καλά και δεν νομίζουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό ως προς την ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι μια καλή λύση, αλλά ίσως δεν πρέπει να την τρεβήξουμε μέχρι τα άκρα. Θα πρέπει να έχουμε μια, ένα τελικό αποτέλεσμα συγκρίσιμο ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε σε σχέση και με την οδηγία για την έγκαιρη προειδοποίηση, τρία χρόνια, περιθώριο που προτείνει η Επιτροπή. Και ναι μεν στην ευελιξία, αλλά δεν πρέπει να χαθούν τα κίνητρα για την αναθεώρηση του στόχου ανακύκλησης μετά από ένα χρόνο. Ναι, σαν βάση, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε τους στόχους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε δηλαδή μετά την εισαγωγή των νέων ορισμών και των μεθόδων υπολογισμού, να δούμε αν τα κράτη έχουν μπορέσει να ορίσουν και να τηρήσουν στόχους. Ένα χρόνο μετά την αναθεώρηση δηλαδή μπορεί αυτό να γίνει. Και εδώ επίσης έχω κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την εισαγωγή της έννοιας προϊόντα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί πρέπει να μπει εδώ ένας ορισμός προϊόν δεν είναι κάτι που πετάμε, δεν είναι κάτι που δεν χρειάζεται πια ο ε, κάτοχός του, άρα δεν μπορούμε να το ταυτίζουμε μετά. τα απόβλητα. Πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική λύση στη διατύπωση, στον ορισμό. Υπολογισμός, μέθοδος υπολογισμού, αν θα έχει αποτελέσματα σωστά. Νομίζω ότι αυτό θα κρυθεί και από τον ε, ορισμό της ολοκλήρωσης διαδικασίας ανακύκλησης και επαναχρησιμοποίησης. Το σημείο υπολογισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνει για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διαδικασία της ανακύκλησης την εισαγωγή νέων προτύπων. Και αν αυτό είναι λογική λύση, δεν ξέρω μήπως είναι και υπερβολική ε, στράτευση στην, ε, στον αγώνα της ανακύκλωσης. Επίσης ένα σύστημα ενημέρωσης και καταγραφής μπορεί να μην είναι πολύ λεπτομερής, αλλά, λεπτομερές, αλλά πάντως χρειάζεται συγκρισιμότητα και για την Επιτροπή. Και πιστεύω θα ήταν καλό να, είμαστε λιγότερο, να είναι λιγότερο εντατική αυτή η παρέμβαση. Η συνάδελφος και επίσης με παρακάλεσε να κάνω μια σύντομη παρουσία στο δικών της θέσεων. Ε, να, το, να μιλήσω τώρα ή να περιμένω να ξανάρθει η σειρά. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Μπούζεκ. Ε, would like to, to, to focus ourselves in the Καλώς πρόεδρος, ε, ας συγκεντρωθούμε στις πρώτες παρεμβάσεις και οδών. Γκίρεκ, S&D. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα στο οποίο πρόκειται να μιλήσω έχει να κάνει με τρεις τύπους αποβλήτων χρησιμοποιημένες μπαταρίες αυτοκινήτων και αντίστοιχα οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Κάθε τύπος μπαταρίας ηλεκτρικής στήλης χρειάζεται διαφορετική χρήση, επεξεργασία και ε, τελικό στάδιο ζωής προϊόντος. Ε, ναι, λοιπόν, είχα το θέμα αυτό. Κοίταξα να δω πού μπορεί να υπήρχαν σημεία συμφόρηση στην οδηγία και μπορούν να βελτιώσουμε τα, την, ε, τις προτάσεις. Σε σχέση με τις ηλεκτρικές στήλες αυτοκινήτων, υπάρχουν ε, κέντρα διάλυσης που προβλέπονται νόμιμα, αλλά υπάρχουν και άτυπα τέτοια κέντρα διάλυσης. Ένα ε, σύστημα γκρίζας αγοράς, θα λέγαμε, με 50% περίπου υπηρεσίες διάλυσης οχημάτων και εκεί πρέπει να πούμε ότι τα μεταχειρισμένα ε, αυτά ανταλλακτικά μπορεί να ξαναπουληθούν και άρα να είναι και επικίνδυνα για την κυκλοφορία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια προσεκτική καταγραφή, να ξέρουμε ποια είναι, πόσα είναι τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στην αγορά και έτσι να μπορούμε να ξαναβρίσκουμε αυτά τα οποία έχουν μείνει σε κυκλοφορία για να έχουμε μια σαφή εικόνα εκείνων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής όμως αυτή η μαύρη αγορά, η άτυπη αγορά δεν επιτρέπει να δούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και πρέπει βέβαια να γνωρίσουμε πότε θεωρείται ένα όχημα ως απόβλητο, από ποια στιγμή θεωρείται υπόβλητο. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λύσουμε σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές και νομίζω έτσι μπορούμε να λύσουμε αυτό το σημείο συμφόρησης. Ε, οι ηλεκτρικές στήλε γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά μολύβδου. Εδώ λοιπόν τεχνολογικά δυσκολία δεν βλέπω, η τεχνολογία μας επιτρέπει την ε, καταργασία τους. Προβλήματα όμως έχουμε για λόγους οικονομικούς. Ο μόλιβδος από την Κίνα είναι τόσο φθηνός ε, πλέον που δεν αξίζει καν τον κόπο η επεξεργασία των στυλών αυτών γιατί δεν αξίζει οικονομικά. Και άρα βλέπουμε πεταμένες ηλεκτρικές στήλες μπαταρίες δηλαδή παντού. Οικιακές συσκευές. Οι λεγόμενες λευκές συσκευές έχουν ε, μεγάλη δυσκολία, χρειάζεται μια διαφορετική λύση, ο τρόπος δηλαδή συλλογής και αποθήκευσης απαιτεί να δοθούν διαφορετικές ε, λύσεις ε, με μια νομική προσέγγιση διαφορετική και κίνητρα ώστε να αποθηκεύονται και να την χάνουν κατεργασίας, περαιτέρω επεξεργασίας αυτές οι συσκευές. Το πρόβλημα εδώ ιδιαίτερος έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία συνήθως αποστέλλονται στην από Ανατολή όπου είναι και φθηνή ενέργεια και δεν είναι τόσο ε, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευαισθησία ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και άρα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο θέμα αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για το πώς μπορούν να ε, διοχετεύονται αυτές οι συσκευέ υπό ποιους όρους και με ποιες διάβλους μπορούν να διοχετεύονται αυτές οι συσκευέ στην ΑΠΟ Ανατολή. Και πρέπει να κοιτάξουμε επίσης και τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Στο ένα και δύο είμαστε ακόμα. Ταντίτσικα. Και Fox. ECR. Σκιώδης. Τελίνσκα, συντάκτης. Κύριος Φόξ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ομάδα μου είναι υπέρ τη οικονομικής αξιοποίηση πόρων ε, και έτσι θα μιλήσω και για τις τέσσερις εκθέσεις εκπροσωπώντας την ομάδα μου. Εκ μέρου των συναδέλφων, ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη δουλειά τους. Διακόπτει ο μίλητης. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετέ επιφυλάξει ως ομάδα για την προσέγγιση που βλέπουμε στην πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή, αλλά και στα σχέδια των εκθέσεων. Θέλουμε μια αναλογική προσέγγιση, η οποία θα εστιάζεται στα κύρια ζητήματα. Η ομάδα μου υποστηρίζει το στόχο της βελτίωση τη διαχείριση των αποβλήτων, τη βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση και ω εκ τούτου και τη. Ε, αξιοποίηση των, ε, της εξοικονόμησης καλύτερα εισαγωμένων ενεργειακών πόρων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μια οικονομική εξέλιξη και δυναμικό που νομίζω όλοι αναγνωρίζουν. Πρέπει λοιπόν να οριστούν ρεαλιστικοί στόχοι και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να είναι υπερβολικά αφενός φιλόδοξοι οι στόχοι ε, και στη συνέχεια και αφετέρου να εξασφαλίζονται παρεκκλήσεις για ορισμένα κράτη-μέλη. Γιατί λοιπόν ορίζονται στόχοι τόσο υψηλοί που δεν μπορεί κανεί να του επιτύχει. Είναι σαν να λέτε ορίζω του στόχου, είναι πολύ υψηλοί, δεν μπορεί να του επιτύχετε, αλλά δεν πειράζει αν αποτύχετε. Να μα εξηγήσει η Επιτροπή λοιπόν γιατί επέλεξε αυτή την προσέγγιση. Δεν θα ήταν καλύτερο να έχει επιλέξει ρεαλιστικού στόχου και να εξασφαλίζει την πλήρωσή του όπω πρέπει. Πώ θα εντοπίζετε σε ποιο κράτο έχει δοθεί η παρέκκληση, όπω στο 11.3 τη οδηγία για τα απόβλητα για τα πρόσθετα μέτρα που προτείνουν οι συγητές και οι συντάκτες δεν είναι ξεκάθαρο με ποιο μέλημα ή πώ έχουν αξιολογηθεί οι συνεπίε του ή αν είναι ε, απαραίτητες οι επιπλέον αυτές προτάσει. προτάσεις. Οι ε, παραδείγματι για τα απόβλητα έλαια με βάση το θεματολόγιο του κανονισμού θα έπρεπε να υπάρχει μια διεξοδική αξιολόγηση συνεπειών για τον καταναλωτή και για τις τοπικές αρχές πριν προχωρήσουμε στην εξέταση μιας τέτοιας πρότασης και θα, έπρεπε να ξέρουμε ότι τα ωφέλη αυτής της πρότασης θα αντιστάθμιζαν την επιβάρυνση ιδιαίτερα για τον ε, κλάδο και μάλιστα τις μικρομεσαίες του επιχειρήσεις. Επίσης ανησυχούμε σε σχέση με τους στόχους, τους πρόσθετους, τους νέους στόχους, τροποποίηση στόχων ε, ενισχυμένη ευθύνη και άλλες αντίστοιχε προτάσεις που έχουν συμπληρωθεί από τους ε, εισηγητές και συντάκτες. Ε, παρακαλώ, μπορέσατε να μετρήσατε αγαπητοί συνάδελφοι τους επιπλέον στόχους που έχετε συμπληρώσει, που έχετε προσθέσει στα κείμενα. Δεν είναι δύσκολο ακόμα και τα θεσμικά όργανα να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την υπόθεση αυτή τους πρόσθετους στόχους δηλαδή και επιβαρύνεται πολύ το σύστημα. Ο κλάδος η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ζητάει εδώ και καιρό πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Σαφείς στόχου, κατανοητούς, που δεν θα αλλάζουν. Κάθε φορά που η Επιτροπή διατυπώνει νέα πρόταση. Η ομάδα μου λοιπόν ανησυχεί ιδιαίτερω και για την πρόταση της Επιτροπής για τι κατεξουδότηση ε, και τις εφαρμοστικές πράξεις οι οποίες μπορούν να σημάνουν σημαντικές αλλαγές για τη βιομηχανική παραγωγή και το κλάδο και έχουμε δει και στο παρελθόν ότι πάντοτε δημιουργούσαν προβλήματα αυτές οι διατάξεις για τις κατεξουδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρεί τον κατάλογο είτε των ε, επικίνδυνων ε, αποβλήτων είτε των πρώτων υλών μόνη της και χωρίς να χρειάζεται να διαβουλευτεί τα κρατη πρέπει να αναλυφθούν ε, μέτρα και να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν ήδη οι μεγάλες μονάδες ε, ανακυκλώνοντας τις πρώτες σύλλες όπου είναι δυνατόν, επειδή τους έχει ζητηθεί. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν ακριβώς την πρόκληση, η οποία είναι τα απόβλητα που παραμένουν πέραν της ανακύκλησης. Πρέπει να δούμε επίσης τις συνέπειες αυτών των προτινομένων διατάξεων, γιατί οι διατάξεις θα επηρεάσουν σημαντικά τμήματα και του ιζουμηχανικής του μηχανικού κλάδου και των τοπικών αρχών, αλλά βέβαια και την πραγματική ζωή των καταναλωτών. Και πρέπει να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των υπερβολικών απαιτήσεων στις φιλοδοξίες και της πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάβορο έχει το λόγο. Μπορείτε να διαχωρίσετε την ομιλία σας γιατί είσαστε εισηγητής και για τις τέσσερις εκθέσεις Μπορεί κάτι να μας πείτε για το, τα, τις εκθέσεις του κυρίου Ταλίτσκα, τις δύο εκθέσεις και μετά στον επόμενο γύρο να λάβετε το λόγο για τις υπόλοιπες δύο. Ευχαριστώ, θα ακολουθήσω τις οδηγίες σας και θα επικεντρωθώ στα, στις ηλεκτρονικές, στα ηλεκτρονικά απόβλητα και την υγειονομική ταφή. Ως προς την υγειονομική ταφή θα ήθελα να πω ότι με τον εισηγητή και του σκιώδης έχουμε κοινό, κοινή αντιμετώπιση της πρότασης της Επιτροπής και υποστηρίζω τη θέση του εισηγητή. Καταρχήν θα πρέπει να πω να μιλήσω για την ξεχωριστή συλλογή βιοποβλήτων που θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και που ανέφερε ο κύριος Φέντερλε που αντικαθιστά τον κύριο Τελίτσκα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει υποχρεωτική η ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Επίσης θα πρέπει να γίνει μία ανταλλαγή πληροφοριών και των ε, πρακτικών για τη χρήση καινοτόμων λύσεων έτσι ώστε να υπάρχει μία συμβίωση στις χωματερές Υπάρχουν ε, πολλές ε, πρωτοβουλίες από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Και σύμφωνο όχι μόνο ως προς την υγειονομική ταφή, αλλά ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να έχουμε μία σωστή βάση δεδομένων και μία κοινή μεθοδολογία καθώς και ορισμούς. Τώρα συζητάμε τα επιμέρους ζητήματα ξεχωριστά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ αυτών και αλληλοστήριξή τους. Μπορούμε να δεχτούμε και διαφορετικούς κανονισμούς που ενδεχομένως αντιβαίνουν ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα συνεκτικό σύστημα. Ως προς την αποστολή αποβλήτων προαναφέρθηκε και σε σχέση και με την υγειονομική ταφή είναι θέμα αυτό, αλλά θα επεκταθώ και ως προς τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Η, η μεταφορά αποβλήτων έχει μεγάλη σημασία γιατί πολλές φορές υπάρχουν και φορολογικές απάτες κατά την αποστολή, γιατί στην ουσία τι κάνουμε, μεταφέρουμε ε, περιβαλλοντικά ε, πόδινα μέτρα και συνέπειες στα νέα κρατημέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι ως προς την υγειονομική ταφή δεν αρκεί να την καταπολεμήσουμε καθεαυτή, γιατί αυτό θα μπορούσε να μην οδηγήσει σε μείωση των αποβλήτων, αλλά να κινηθούμε προς την αποτέφρωση που δεν είναι στόχος του πακέτου κυκλικής οικονομίας. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια κατά την καταπολέμηση της υγειονομικής ταφής και να δημιουργήσουμε νέους ε, στόχους χωρίς να υπάρξει αποτέφρωση ως προς τις ε, μπαταρίες και τους ισορρευτές τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και εναρμονισμένη μεθοδολογία καθώς και ορισμούς σε σχέση με τις μπαταρίες και τους σωρευτές ε, ως προς την αποστολή των αποβλήτων. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός. Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστούμε πολύ αυστηρά, έτσι ώστε να μην γίνουν αποστολές αποβλήτων χωρίς να ελέγχονται. Τέλος, ε, το παράρτημα ίσως θα πρέπει να καταρτιστεί περισσότερο για να λάβουμε υπόψη όλες τις συνιστώσεις του πακέτου σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων και τη μεταφορά τους και μέσα στα πλαίσια της οδηγίας πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλικιώτης, παρακαλώ. Αν θέλετε να χωρίσετε την ομιλία σας, πρώτα να μιλήσετε για τους δύο φακέλους και μετά για τα υπόλοιπα, σε ένα δεύτερο γύρο. Για το τρίτο και το τέταρτο, όπως θέλετε. Αν θέλετε και τα τέσσερα μαζί, όπως θέλετε εσείς. Είναι στη διακριτική της Ε, επειδή δεν έχω χρόνο, θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω μόνο για την ε, τροποποίηση της οδηγίας για τα απόβλητα. Ε, και στην ατζέντα μας ήταν αυτό το θέμα ως πρώτο, ως ε, θέμα 11 και θα μιλήσω μόνο γι' αυτό ε, στο οποίο είμαι και σκιώδης συγκητής. Ε, δηλαδή θα μιλήσω για την ε, αναθεωρημένη οδηγία για τα απόβλητα. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον, τον συνάδελφο τον Μύρο Σλατοπόσε, που έχει επιτύχει με τη δουλειά του να προ, προ, προτάξει βελτιώσει στην πρόταση της Κομισιό. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά θεωρούμε ότι πρέπει αυτή η αναθεωρημένη οδηγία να συμβάλλει καθοριστικά στη συνετή και ορθολογιστική χρήση των πόρων, καθώ και στη μείωση τη παραγωγή αποβλήτων, με στόχο βεβαίω την προστασία του περιβάλλοντο και τη υγεία των ανθρώπων, για βελτίωση τη ποιότητα τη ζωή μα. Ε, πρέπει να γίνουν ε, πάρα πολλά προ ε, υλοποίηση αυτού του στόχου. για μα αρχικά είναι σημαντικό να ενισχυθεί η πρόληψη με ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στην ανακύκλωση. Ε, εξίσου σημαντικό είναι να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι, δηλαδή να τονιστεί η ευθύνη των μεγάλων παραγωγών, να αναπτυχθούν δημόσιες υποδομές, να ενισχυθεί ο δημόσιος έλεγχος, να ευθαρρυνθεί η χρήση μέσων που περιορίζουν την περιβαλλοντική ρήπαση, ε, να ευθαρρυνθεί η επεξεργασία ρημάτων με σκοπό την παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρική ενέργεια, να προωθούν μέτρα για κατάλληλη υγειονομική ταφή των αποβλήτων και μέτρα βεβαίω για αποκατάσταση τη γη, ιδιαίτερα εκεί, που γίνονται ταφές. ταφέ. Στη διαδικασία διαμόρφωση νομοθεσία είναι πολύ σημαντική συμμετοχή των τοπικών αρχών, των κοινοτήτων, καθώ βεβαίω και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εμείς θεωρούμε πολύ θετικά α, ε, τα νέα στοιχεία που προσθέτει ο συγητής όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παραγωγών, την ανάγκη ενίσχυση των δικαιωμάτων ε, των καταναλωτών, ε, για παράδειγμα η διασφάλιση δωρεάν πρόσβαση σε αισθήματα συλλογής και ανακύκλωσης, καθώς και η, η πρόταση για ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ορυκτέλεων και των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι πως δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τις ίδιες δυνατότητες, ούτε βρίσκονται στο ίδιο σημείο εκκίνησης, ώστε να μπορέσουν να ελοπίσουν τους νέους στόχους που θα τεθούν. Ιδιαίτερα, τα κράτη που έχουν πληγεί από τις νεοφιλελεύθερες, τις μνημονιακές πολιτικές της σκληριδότητας, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ε, σε μια φοβερή κρίση και φτωχοποίηση του λαού. Άρα είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν κονδύλια από τα διαφθορτικά και τα επενδυτικά ταμεία της Ένωσης για να χρηματοδοτηθούν τα κράτη, αυτά ώστε η ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται για τη διαχείριση των αποβλήτων, για την ανακύκλωση, να μπορούν να, να, να, να υλοποιήσουν αυτές τις υποδομές, όπως βεβαίως και τις αποζημίες που, που δικαιούνται και πρέπει να καταβάλουν στις κοινότητες, στον χώρο τον οποίο βρίσκονται οι χώροι υγειονομικής ταφής, και είναι προς αυτήν την κατεύθυνση που θα καταθέσουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο δεύτερος γύρος. Τέσσερις ομιλητές έχω, σκιώδες συγητές. Η κυρία Βίρκουνεν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα πράγματα έχω να πω για τα ηλεκτρικά απόβλητα, τους σωρευτές, μπαταρίες και το τέλος ζωής. Η πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μικρή και αφορά μόνο την αναφορά στατιστικών στοιχείων και βεβαίως το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ε, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα για να έχουμε και στόχους ρεαλιστικούς για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε σήμερα για να έχουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για το μέλλον. Από τα σημαντικότερα λοιπόν ποιο είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους και να ε, κοινοποιούν τα ίδια στοιχεία και αποτελέσματα των μετρήσεων για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε όπως πρότεινε άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση Τελίτσκα είναι καλή, οι προτάσεις επίσης και θέλω να τον ευχαριστήσω για την δουλειά του το ΕΛΚ μπορεί να υποστηρίξει τα περισσότερα από όσα προτείνει ο εισηγητής. Όπως είπε και ο ίδιος, έχει σημασία να έχουμε ίσους όρους παιχνιδιού μεταξύ των διαφόρων φορέων της αγοράς για να έχουμε σωστή διαχείριση των αποβλήτων για λύσεις υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ της αγοράς και φθηνές. Προτείνει διάφορα οικονομικά μέσα και εργαλεία και για τις τρεις οδηγίες ο εισηγητής. Βασικός στόχος είναι να μεταφερθούμε προς μια κυκλική οικονομία και είναι σωστή αυτή η φιλοσοφία. Έχει σημασία οι επιχειρήσεις να έχουν κίνητρα για να προχωρούν στη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά θα πρέπει πολύ προσεκτικά ε, να ε, δούμε τι χρήση θα κάνουμε ποιών εργαλείων με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Χρειάζεται ακόμα συζήτηση το θέμα αυτό ε, σε απότερο στάδιο συμφωνεί το ΕΛΚ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να απλουστεύεται ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούνται από τα κράτη-μέλη ε, τα στοιχεία αυτά για να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία. Επίσης πολύ καλά κάνει ο εισηγητής και τονίζει ότι υπάρχουν προβλήματα ε, στη διαχείριση και στην επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Είναι σημαντικό όλα τα ε, απόβλητα αυτά που ε, ε, διαλέγονται και συλλέγονται ξεχωριστά να την χάνουν και τη σωστή επεξεργασία. Αλλιώ τι να την κάνουμε τη διαλογή και τη χωριστή συλλογή. Η ανακύκλωση είναι που κάνει τη διαφορά. Αυτά από πλευρά του ΕΛΚΑ και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Η κυρία ε, Κατλίν ε, Φανμπρέμπτ ε, αντικαθιστά την κυρία Μούντι που είναι μάλλον εκεί στις Βρετανίες. Ναι, έχει πολλή δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εποχή ε, και ελπίζω να κάνουν καλή δουλειά και να κερδίσουν το δημοψήφισμα. Λοιπόν, σύντομα να σας πω τι λέει η κυρία Μούντι. Είναι σκιώδη συγγήτρια για την οδηγία για τα απόβλητα των ε, συσκευασιών και της συσκευασίας. Ε, um, ε, ε θέλουμε να εθαρρύνουμε την επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας φυσικά, ε, γιατί Ε, μπορεί ε, η ε, επέκταση της ευθύνης του κατασκευαστή να οδηγήσει στην παραγωγή νέων πρώτων υλών, αλλά δεν θα έχουμε αγορά για να τα απορροφήσει. Κυρίως αυτό αφορά τα πλαστικά και τα μπουκάλια. Οι γυάλινες φιάλες δηλαδή. Για να ε, λειτουργήσουν όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα ε, για τους παραγωγούς έτσι ώστε οι συσκευασίε που παράγουν να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και να είναι και πιο βιώσιμες. Ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα τα χρώματα ε, στα πλαστικά. Είναι πολύ δύσκολο μια πλαστική συσκευασία να ανακυκλωθεί όταν είναι πολύχρωμη. Άρα ε, θα πρέπει να δίνονται ανάλογα κίνητρα για να χρησιμοποιούνται λιγότερα χρώματα. Αντίστοιχα ισχύουν και για τις γυάλινες συσκευασίες. Η συμπεριφορά του καταναλωτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό θα ζητήσουμε ε, ένα νέο είδος επισήμασης, νέα ε, μορφή ε, προβολής όλων αυτών των ε, συσκευασιών και με ένα σήμα, μια σφραγίδα που όλα αυτά να τα προωθεί και να τα επιβραβεύει. Στη θάλασσα έχουμε πρόβλημα, ξέρετε ότι κινδυνεύουν τα θαλάσσια θηλαστικά και θα πρέπει να έχουμε και στόχους φιλόδοξους αλλά και δεσμευτικούς για να μειώνονται τα απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα. Ανησυχούμε πάρα πολύ. για την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών. Μπορεί να ανακυκλώνουμε, αλλά συνήθως αυτά είναι μίας χρήσης και πετιούνται τα ανακυκλωμένα. Άρα εκεί θα χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Κυρία Ζαμπόρσκα. Είναι σκιώδης επίσης και από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Την αντικαθιστά ο κύριος Ρόιλ. Παρακαλώ. Ναι, και εγώ ένα χαρτάκι πήρα. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω. Δυστυχώς σήμερα κολλείεται. Δεν συμφωνώ μαζί της σε όλα τα σημεία, αλλά πάντως αυτή είναι η συζήτηση. Λοιπόν, για την αποφυγή των αποβλήτων, ε, οι δείκτες ε, των κρατών μελών, θα πρέπει να εισάγονται στα εκάστοτε προγράμματα αποφύγης αποβλήτων και πρέπει να προστίθενται, λέει η κυρία Ζαμπόρσκα και τα σχετικά κίνητρα για την αποτέφραωση. Δεν πρέπει να ενισχύεται κανένα σύστημα αποτέφρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι πιο αυστηρές διατάξεις, ε, σαφείς ε, διατάξεις για την απόθεση και την αποτέφρωση, αποτέφρωση, ποτέ αποτέφρωση βιολογικών αποβλήτων. Βιολογικά απόβλητα χρειάζονται ένα επιπλέον ευρωπαϊκό στόχο. Εγώ είμαι κάπως πιο επιφυλακτικός εν προκειμένου. Θαλάσσια απόβλητα να περιληφθούν μας λέει η κυρία Ζαμπόρσκα επίσης, ευθύνη παραγωγού, θετικά. συγκεκριμένες προτάσεις διατυπώνει για τα εθνικά προγράμματα, υποστηρίζει τις, τα εθελοντικά εθνικά προγράμματα δράσης η κυρία Ζαμπόρσκα, όπου θα πρέπει να περιγράφεται και ο τρόπος επίτευξης των προσδοριζομένων στόχων και ε, ζητάει να προτιθούν νέοι ορισμοί και αυτά ήταν εν ολίγης οι σύντομες παρατηρήσεις κυρία Ζαμπόρσκα για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συγκεκριμένε παρατηρήσει της Μαντάμ Ζαμπόρσκα. Γιάβορ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με τρεις πιο γενικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, όταν η Επιτροπή απέρριψε την δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, το είχε πράξει επιχειρηματολογώντας πως το επόμενο σύνολο προτάσεων θα ήταν πολύ πιο φιλόδοξο και σε σχέση με την κυκλική, με την αποτελεσματικότητα στην κυκλική οικονομία, αλλά αυτό δεν απεδείχθη στην πράξη, καθώς η πρόταση που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο Επιτροπή δεν είναι πιο φιλόδοξη από ό,τι η προηγουμένη, είναι του αντίον λιγότερο φιλόδοξη και μάλιστα δεν καλύπτει καν την ε, παραγωγή, τον κλάδο της παραγωγής. Λυπούμε λοιπόν ιδιαίτερως που δεν ήταν αληθής η επιχειρηματολογία της Επιτροπής. Πρώτη και γενική παρατήρηση και επίσης ανέφερα ήδη πως μιλούμε για τέσσερα ανεξάρτητα μεταξύ τους θέματα, ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει η συνοχή, η συνεκτικότητα των τεσσάρων αυτών ε, πακέτων και να μην ε, διατυπωθούν δικαρονιστικά κείμενα τα οποία θα είναι μεταξύ τους αντιφατικά. Περιβάλλον ή καλύτερα ρεαλιστικοί στόχοι αντίθετα από τις θέσεις του ECR. Εμείς οι πράσινοι πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους και εφικτούς. Στόχους που θα επιτυγχάνονται με συνεργασία κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να προσδορίσουμε και να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους. Για την οδηγία πλαίσιο πρέπει να αναφέρω ότι λυπούμε ιδιαίτερος για το δεν αναφέρονται στόχοι για τα απόβλητα τροφίμων και τα θαλάσσια απόβλητα. Εγώ θα προτείνω 50% μείωση για τα απόβλητα τροφίμων και τα θαλάσσια απόβλητα ε, είναι τεράστιο το πρόβλημα, είναι φρικτό το πρόβλημα και επίσης θα ήθελα περισσότερη προσοχή να δοθεί στο εμπορικό και βιομηχανικό, στα ε, εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα, γιατί μιλούμε συνήθω για δημοτικά απόβλητα, αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη τα εμπορικά και τα βιομηχανικά. Τα γεωργικά επίσης τα έχουμε ξεχάσει τελείως και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι σημαντικός όγκος αποβλήτων, τεράστιος όγκος αποβλήτων που θα πρέπει να ε, την χάνουν ε, διαχείρισης ε, κατάλληλης. Επίσης, οι επικίνδυνες ουσίες στα απόβλητα. Η ανακυκλισμότητα των αποβλήτων ξέρουμε ότι εξαρτάται από το εάν υπάρχουν επικίνδυνε ουσίε ή όχι. Γιατί αν υπάρχουν επικίνδυνε ουσίε είναι πολύ δύσκολη η ανακύκλωση. Άρα θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία ε, της ύπαρξης φιλόδοκων στόχων για κομποστοποίηση 65% έως το 2025 ε, που έχουμε ήδη αναφέρει, πιο φιλόδοξη προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση γιατί αποτελεί τη βάση κάθε κυκλικής οικονομίας. Επίσης, η χρήση χώρων απόθεσης χωματερών ε, θα πρέπει να ε, παραταθεί ίσως, αλλά δεν πρέπει να αναμειχθεί με την αποτέφρωση. Στις συσκευασίε και απόβλητα από συσκευασίε και πάλι, όπως αναφέρθηκε, από τον εισηγητή κύριο Φερέιρα, χρειαζόμαστε σαφή και συνεπή ορισμό φιλόδοξους ε, στόχους ανακύκλωσης ε, συσκευασιών κατά 80% στο 2030, αντίστοιχη με αυτή της ε, πρότασης για την κυκλική οικονομία της προηγούμενης ε, σύνθεσης Επιτροπής και δεν συμφωνώ με τον ορισμό της προετοιμασίας για να επαναχρησιμοποιήσει γιατί μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και χρειάζονται συστήματα προαγωγής της επαναχρησιμοποίησης στον κύκλο των αποβλήτων από συσκευασία. Εναρμονισμένα συστήματα σε όλη την Ευρώπη με συνεκτική σήμανση, επισήμανση αποβλήτων εναρμονισμένη σε όλη την Ευρώπη, στο ο καταναλωτή να μπορεί να καταλαβαίνει πώ λειτουργεί το σύστημα τη επισήμανση αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μποναφέ. Η κυρία Σιμώνα Μποναφέ ας ε, μας πει ποια είναι η άποψη της ΕΜΒΗ. Είσαστε υπεύθυνοι και για τις τέσσερις γνωμοδοτήσεις και γι' αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι μια πολύ σημαντική δυνατότητα που μου δίνετε εδώ, γιατί αύριο θα συζητήσουμε ολόκληρο το πακέτο στην ΕΝΒΗ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ολόκληρο πακέτο και για τις τέσσερις οδηγίες. Και όχι μόνο για την εισηγήτρια και για τις τέσσερις οδηγίες, αλλά επειδή νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με τέσσερις διαφορετικές προτάσεις που αφορούν την πολιτική μας για τα απόβλητα. Όμως θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν αφορά μία ε, πολιτική περιβάλλοντος ή διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά μιλάμε για την επιβολή ενός νέου βιώσιμου βιομηχανικού μοντέλου και για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και φυσικά μπορούμε να προβάλλουμε επιπτώσεις και στην ανταγωνιστικότητά μας. Ξέρουμε ότι είμαστε πολύ φτωχοί σε πρώτες ύλες που ενέχουν ένα πολύ υψηλό κόστος και γι' αυτό πιστεύω ότι από την ανακύκλωση και ανάκτηση υλών μπορούμε να βοηθήσουμε και την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι συνεισφέρει Φέρατε όλοι οι συγητές και σκιώδεις και φυσικά θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση. Τώρα, επί της ουσίας, ε, ε, επί της ουσίας μιλώντας ε, ως προς τους στόχους, είδα ότι ως προς την υγειονομική ταφή και τους στόχους ανακύκλωσης, Καθώ καθώς και τους στόχους συσκευασίας έχουμε αποκατάσταση της αρχικής πρότασης της Κομισιόν που εγκρίναμε με μεγάλη ε, πλειοψηφία στην έκθεση Πίτικάινεν πέρσι. Πρόκειται για στόχους που λαμβάνουν υπόψη φιλοδοξίες αλλά και μία πραγματιστική προσέγγιση, γιατί είναι στόχοι στους οποίους έχουν φτάσει ορισμένα κράτη-μέλη, που σημαίνει ότι είναι εφικτοί. Βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με, διαφορετικές, ε, με 28 διαφορετικές πραγματικότητες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κατεβάσουμε τον πύχη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη που έχουν καθυστερήσει να φτάσουν στους στόχους αυτούς. Μέσω της στοχοθέτησης των διαρθρωτικών ταμείων για την κυκλική οικονομία και επειδή ο χρόνος παίζει μεγάλο ρόλο, ο Επίτροπος Κατάινεν στην προηγούμενη Ολομέλεια μας είπε ότι και το σχέδιο Γιούνκερ θα χρηματοδοτήσει την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό νομίζω ότι φέρουμε ευθύνη και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να φτάσουμε σε ένα σαφές σύστημα κανόνων έτσι ώστε και οι επενδυτές να μπορέσουν να κάνουν το δικό τους υπολογισμό. Έχουμε να κάνουμε με νέα βιομηχανικά πρότυπα. Και γι' αυτό οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αν μιλάμε για στοχοθέτηση, δεν σημαίνει ότι θα βασιστούμε μόνο σε αυτήν. Το πρώτο βασικό βήμα είναι αυτό της πρόληψης ε, συσσόρευσης αποβλήτων μέσα πλαίσια αυτής της ιεράρχησης διαχείρισης αποβλήτων από την πρόταση της Κομισιόν και τη δική μας πρόταση και εισηγητών της ΕΜΒΗ. Μιλάμε για ε, μία συσκευασία αποκλειστικής χρήσης, μοναδικής και αποκλειστικής χρήσης και αυτή την οδηγία θα τη δούμε. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να αποκλείσουμε ή να μειώσουμε την παραγωγή αποβλήτων, διότι προβάλλουμε όλους τους ε, μηχανισμούς καινοτομίας για να έχουμε μια απλούστερη συσκευασία, προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να ε, ανακυκλωθούν έτσι ώστε να γίνεται μία χρήση προς τα άνω. Καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι αυτό το πακέτο. Ένα άλλο θέμα ύψης της ε, σημασίας της κυκλικής οικονομίας αφορά τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, δηλαδή να ορίσουμε οικονομικά μέσα και να απλουστεύσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες που κινούνται στη, προς την βιομηχανική συνδύωση. Δηλαδή, μέσα στα πλαίσια της απλούστευσης της διαχείρισης των αποβλήτων, χωρίς να υπάρξουν στρεβλώς στην ενιαία αγορά. Πρόκειται για σημεία που συμμερίζομαι. Ναι. Έχω μία μόνο αντίρρηση Μιλήσαμε για μεθόδους υπολογισμού για την ανακύκλωση. Θα πρέπει να έχουμε μια εναρμονισμένη μέθοδο υπολογισμού. Διαφορετικά θα φτάσουμε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επίσης, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αστικά απόβλητα και τελειώνω πρόεδρε γιατί μιλάμε για το 7% των αποβλήτων τα αστικά απόβλητα είναι μόνο το 7% των συνολικών αποβλήτων. Γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα, όχι για να βάλουμε για άλλους, να θέσουμε άλλους κανόνες στις βιομηχανίες, αλλά για να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πρώτες ύλες. Πρόκειται για μια περίπλοκη φιλοδοξία, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το στίχημα. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία μου για τα σχόλιά σας. Ελπίζω ορισμένοι από τους συγητές και τους κοιόδες να είναι παρόντες αύριο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και τώρα θα παρακαλούσα ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Είναι ο κ. Βίλιος Λάγκενορφ Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνετε μερικά λεπτά. Προφανώς στο παρόν στάδιο και το ίδιο ισχύει και για αύριο είμαστε στη φάση της ακρόασης, δηλαδή ακούμε ε, τις δικές σας προτάσεις και τα σχόλια και θα είμαστε σε πολύ στενή επαφή ε, τους επόμενους μήνες. Τούτων λεχθέντων όμως Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το σχέδιο εκθέσεις των τεσσάρων συντακτών γνωμοδότησής σας. Είναι σαφές ότι υποστηρίζετε γενικά την κατεύθυνση που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας χαροποιεί αυτό. Θεωρείται θετικά αυτά που προτείνουμε για την καλύτερη διαχείριση και την ιεράρχηση ως ένα ε, θετικό για την κυκλική οικονομία, όχι το αποκλειστικό στοιχείο και αναγνωρίζετε ότι και οι στόχοι και τα εργαλεία πολιτικής και οικονομικής και άλλης έχουν σαφή ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή τη διαδικασία και την πορεία. Βεβαίως, αν δούμε τους στόχους πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις σχετικά με το ποιους στόχους θέλουμε, για ποια απόβλητα, ποια θα πρέπει να έχουν στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μήπως είναι καλύτερο να έχουμε εθνικούς στόχους και επίσης σε ποιο επίπεδο και πώς θα οριστούν οι στόχοι αυτοί. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα ε, για το τι εννοώ. Στην πρότασή μας, ε, το έχουμε ξανασυζητήσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά τα αστικά απόβλητα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η στόχη μας πάρα πολύ φιλόδοξη. 65% είναι ο στόχος ανακύκλωση για το 2030. Είναι πολύ φιλόδοξος για τα αστικά απόβλητα, αλλά θα πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα στα κράτη-μέλη ε, γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει εδώ μια ρήτρα αναθεώρησης προς τα πάνω το 2025 για να φτάσουμε και στο 70% αν θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ότι έχουν κάνει πρόοδο τα κράτη μέχρι τότε. Άρα αναλύουμε την ανάλυση αυτή και έχουμε υποστηρικτικό ε, ρόλο στη μελέτη αντικτύπου. Τώρα, για τους νέους στόχους θα πρέπει πάντα να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση, ποιες είναι οι συνέπειες ε, αυτών που ζητούμε. Για παράδειγμα, στόχοι που προτείνονται για τα ορυκτέλεα και τα άλλα χρησιμοποιημένα ελέα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιο στόχο ε, αριθμητικό χωρίς να έχει γίνει η σωστή ανάλυση. Το ίδιο ισχύει για τους ευρωπαϊκούς, πανευρωπαϊκούς στόχους. Χρειάζεται ανάλυση πολύ καλή, όπως προτείνει η έκθεση άλλωστε. Και εμείς το προτείναμε. Σε σχέση με τα βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα. Ε, θα πρέπει να γίνει λοιπόν πάντα μια πολύ καλή καταγραφή της ε, πραγματικότητας που ισχύει στα κρατημέλη πριν προτείνουμε στόχους ανακύκλωσης για τα εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα. Έτσι θα πρέπει να θέτουμε στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό εξηγεί ε, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στόχος για τα απόβλητα τροφίμων, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τη μεθοδολογία πριν ορίσουμε τέτοιους στόχους, πώς θα γίνει αυτό. Αυτό φαίνεται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαφέστατα. Πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή και ποιο είναι ο ορισμό για τα απόβλητα τροφίμων πριν συνεχίσουμε στη μεθοδολογία. Ε, Είμαστε προσεκτικοί λοιπόν προς το παρόν. Με χαρά να δούμε και περαιτέρω και πιο φιλόδοξους στόχους. Θα έχουμε χρόνο να το κάνουμε, όμως χρειάζεται ανάλυση της παρούσας κατάστασης και μελέτη αντικτύπου πριν προχωρήσουμε. Έρχομαι τώρα σε μερικά από τα μέσα και εργαλεία που προτείνουμε. Βλέπουμε μεγάλη υποστήριξη για κάτι που ζητάει η πρόταση ε, μέσα οικονομικά μέσα συνοδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Στο σημείο 4 το προβλέπουμε. Αιτιολογική σκέψη 7 που απαριθμεί ε, διάφορα οικονομικά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο κύριος Τέλιτσκα πρότεινε στα παραρτήματα για τις μεμονωμένες οδηγίες. Νομίζω καλύτερο είναι να γίνει αυτό στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα που είναι κεντρική παρά στις επιμέρους ε, τομεακές αν θέλετε. ότι θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα, δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Το γράφει η πρότασή μας. Για το EPR έχουμε κάνει προτάσεις για τις γενικές απαιτήσεις. Ας πούμε, η ανάκτηση, η κάλυψη η πλήρης του κόστους ή όλου του κόστους, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν το έχουμε ορίσει και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται αυτά ε, τα ε, συστήματα. Ε, στις μπαταρίες σήμερα υπάρχει και σε άλλα είδη υποχρέωση. Δεν ξέρω και κατά πόσο θα πρέπει να επεκταθεί και για τις ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό ακόμα δεν έχει επιληθεί. Επίσης, να πω τώρα και κάτι που μας ανησυχεί και έχει να κάνει κυρίως για την επισήμανση. Το EPR είναι η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Τώρα, για τους στόχους, για την επισήμανση και γενικότερα για τους στόχους, υπάρχει έδαφος για ανησυχία, διότι αυτό που προτείνουμε εδώ είναι στο βαθμό που δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους της ανακύκλωσης, αποτεφρώνονται όλα τα σκουπίδια για παραγωγή ενέργειας, αυτό υπονομεύει την ιεράρχησή τους. Δεν θέλουμε παρατάσεις για αυτό το σύστημα, για τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν φτάσει στο στόχο ανάκτηση και ανακύκλωση των συσκευασιών τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Και μια άλλη ανησυχία, τελειώνω, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ σωστή ισορροπία ανάμεσα στους στόχους τους περιβαλλοντικούς και τους εμπορικούς για την αγορά δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε το όσο ορίζει το άρθρο 18 και να είμαστε προσεκτικοί γιατί η οδηγία για τις συσκευασίε ε, έχει μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία. Αυτό φαίνεται και από την νομική βάση που έχει επιλεγεί. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφοι Πόχε και Φερέιρα για τα τελευταία σχόλια. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που τροποποιεί την οδηγία και που θα ενσωματωθεί στην οδηγία αργότερα πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης για να μεταβούμε σε μια κυκλική οικονομία. Ορισμένες πτυχές αυτής της γνωμοδότησης θα πρέπει να διευκρινιστούν έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια για τη, με την οδηγία για τα αποβλήτα, δηλαδή να δούμε τις συνέργειες και να υπάρξει και ένας αλληλένδετος χαρακτήρας με τους στόχους, να δούμε τα οικονομικά μέσα, πώς να τα υποστηρίξουμε και να τα συμπληρώσουμε. Επίσης θα θέλαμε να δούμε και την πολιτική μας για την πρόληψη των αποβλήτων μέσα στα πλαίσια της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι σκιώδεις θα συνεδριάσουν στο Στρασβούργο τον Ιούλιο και θα ήθελα να ασχοληθούμε με, αυτές, με αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που συνεισέφεραν στη συζήτηση και θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να συνεργαστώ με τους σκιώδεις και όλους τους ενδιαφερόμενους στο εγγύς μέλλον. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω πολύ σύντομα σε σχέση με τους στόχους, αν είναι ρεαλιστικοί, αν είναι υπερβολικά φιλόδοξοι. Για να προβούμε λοιπόν σε μια αποτίμηση θα πρέπει να αναλύσουμε τους στόχους κάθε αυτούς αλλά και τις προθεσμίες. Την προθεσμία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν έχει νόημα να ορίσουμε έναν στόχο που αύριο ε, δεν θα είναι εφικτός. αναγνωρίσουμε τη μεγάλη, ε, τη διαφορετική προσέγγιση των κρατών μελών, γιατί για ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν δυσκολίες ε, για να εκπληρώσουν τους στόχους, αλλά κράτη όμως έχουν δυσκολίες. Για ορισμένα κράτη είναι μεγάλες οι δυσκολίες, για άλλα μικρότερες. Η συνάδελφος Μποναφέ μίλησε για αυτή τη διαφορετικότητα και είπε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς που βρίσκονται μακριά από τους στόχους. Το ζήτημα όμως αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη ε, σοβαρά. Φυσικά θα πρέπει να γίνει πολύ καλή χρήση των διαρθρωτικών ε, ταμείων. Αλλά αυτό το είχαμε δει και πριν με τη χρήση του σχεδίου ε, Juncker. Βρισκόμαστε όμως στο, στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που κάνουν πολύ χαμηλή χρήση. Δηλαδή πολλά κράτη-μέλη ε, δεν χρησιμοποιούν αυτό το μέσον. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε στόχους με νέα μέσα για την επίτευξή τους. Δεν μπορούμε να ορίσουμε νέους στόχους με τα παλαιά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό με την πρότασή μου προσπάθησα να χρησιμοποιήσουμε το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή τις προθεσμίες. Δηλαδή για αυτούς που έχουν ε, μεγαλύτερες δυσκολίες δεν θα φτάσουν σε αυτούς τους στόχους αύριο, αλλά μεθαύριο. Δηλαδή δεν αποδυναμώνουμε τους στόχους, τους δεχόμαστε, αλλά λέμε ότι σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει κανείς λίγο αργότερα σε αυτούς τους στόχους. Υποαιρέσεις βεβαίως καταρχή να υπάρχει μία πορεία βαθμιαίας προσέγγισης από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο άφηξη, θα πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία προσέγγισης, προοδευτικής προσέγγισης. αυτή είναι μια συνθήκη, ένας όρος για να μην υπάρξουν λαθροχειρίες και κολυσιεργίες. Γνωρίζουμε όμως ότι η πορεία αυτή θα είναι λίγο διαφορετική. Και φυσικά θα υπάρχει και η χρήση αυτού του νέου μέσου, δηλαδή της έγκαιρης προειδοποίησης. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντάξουν αυτούς τους στόχους ε, σε αυτή την πορεία προοδευτικής σύγκλησης. Δεν δέχομαι την άποψη της Επιτροπής απόλυτα. Δεν υπάρχει λόγος για τόσο μεγάλη ανησυχία. Θα πρέπει να υπάρχει επανισορρόπηση μεταξύ, του στόχου, μεταξύ των στόχων της αγοράς και του περιβάλλοντος και αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε και στους δύο πόλους χωρίς να αμφισβητήσουμε κανέναν και να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα θετικά προηγούμενα που υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, σας ευχαριστώ για τη σκληρή σας εργασία και σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας εδώ, για την υπομονή σας, γιατί δεν είμαστε πολλοί μέχρι το τέλος των ε, εργασιών μας. Στις 3 η ώρα το απόγευμα θα τα πούμε, η κυρία Μπιελκόφσκα, θα έρθει εδώ η Επίτροπος, η κυρία Μπιελκόφσκα και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 16η Ιουνίου 12 το μεσημέρι. 16 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας για δυόμιση ώρες. Θα τα πούμε στις 3. Γεια σας.